και θα υποβάλουμε αύριο ή στους συναδέλφους θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Αύριο θα ψηφίσουμε και προχωρούμε τώρα και παρακολουθούμε το επόμενο θέμα, την έκθεση ε, του Κλοντ Μοράες ε, σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής οδηγίας 2003 κάθετος 109 ΕΚ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Καταρχήν θα ήθελα ε, να δώσω το λόγο εις ε, τον κύριο Μωράη, συζητητή, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ φοβάμαι διότι όσο φτάνω στην πρώτη παράγραφο θα μείνουμε ελάχιστη συνέθουσα. Με συγχωρείτε, ε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από το συντονιστή του ΕΛΚ, αλλά ευχαριστώ το συντονιστή του ΕΛΚ που παρέμεινε εδώ και με περιμένει τέτοια ώρα νυχτιάτικα. Θέλω να ευχαριστήσω κύριε κυρία Επίτροπε εσάς προσωπικά για την εξαιρετική ε, εργασία που κάνατε να περισσώσετε μία πρόταση η οποία τώρα ε, μπορεί να ε, καλύψει αυτούς που δεν έπρεπε ποτέ να έχουν αποκλειστεί από την οδηγία για την μακροχρόνια διαμονή και με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνουμε αυτή την ατέλεια AUTHORWAVE υπάρχει η, πρόταση της Μαρτίν Ρορ της ε, προηγούμενης εισηγήτριας ε, και θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες και το Συμβούλιο και όποιος δεν ήταν προηγουμένως εδώ θέλω να πω ότι ευχαριστώ όλους και χάρη στη Βελγική Προεδρία μπορέσαμε να προχωρήσουμε και είμαι πολύ ευγνώμων. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει όλους ε, οι οποίοι παραμένουν για πέραν των 5 ετών να μπορέσουν να ρυθμιστούν και τουλάχιστον θα δώσει τέλος στην ανασφάλεια η οποία υπήρχε ε, στο καθεστώς των επιμακρών διαμενόντων ως προς την έκβαση της προστασίας τους. Βέβαια ε, στηρίξαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το να επιτευχθεί ο χρόνος αυτός των 5 ετών ε, και δυστυχώς δεν συνεφώνησε το Συμβούλιο και ορισμένα κράτη-μέλη. Η συμβιβαστική λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων ήταν ότι θα ληφθεί υπόψη η μισή διαδικασία και αν η διαδικασία ξεπεράσει τους 18 μήνες τότε θα ληφθεί πάλι υπόψη. Δυστυχώς πρέπει να επανέλθω στους πίνακες συσχετισμού και πρέπει να τους σχολιάσω παρόλο που θα προτιμούσα να το αποφύγω. Δηλαδή, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιλύσει οριζόντια την κατάσταση αυτή και να αναγνωρίσει τη σημασία των πινάκων συσχετισμού για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα διάφορα νομοθετήματα. Πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό θα δέχεται να καθυστερούσε την όλη διεκπαιρέωση του θέματος και γι' αυτό όσον αφορά την επικουρική προστασία νομίζω ότι πρέπει να ευθυγραμμίσουμε την προστασία μας εις ε, τις προηγούμενες οδηγίες και ε, θα πρέπει τώρα όσοι εποφελούνται από αυτή την οδηγία να γνωρίζουν ότι η προστασία ε, δεν είναι ένα θέμα το οποίο να εγκαταλείπουμε ποτέ και θα χρειάζεται σε περίπτωση απελάς εκπρόσεως από ένα κράτος μέλος να ληφθεί υπόψη και η γνώμη του κράτους το οποίο έχει προσφέρει την προστασία θα πρέπει συγχρόνως να υπάρχουν ε, οι εθνικές ρυθμίσεις κατά τρόπον ώστε ε, να ε, αποφύγουμε την απομάκρυνση και είναι σαφές ότι στις περιπτώσεις που δεν θα είναι προς όφελος των κρατών μελών να ακολουθήσουν το άτομο το οποίο να απελάβνεται δεν θα είναι αυτόματη η απέλαση και τις οικογένειας αφορά το άσυλο και την ε, νόμιμη ε, ε, με την μετανάστευση ε, θέλουμε να μπορέσουν τα θέματα αυτά να καλυφθούν από την νομοθεσία θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, σκιώδεις εισηγητές και τους συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν εις την επίτευξη αυτής της συμφωνίας και της ευχάριστης τριμερούς συνδιαλλαγής αν αυτό δεν αποτελεί παρανόηση. Ευχαριστώ κύριε βουλευτά και τώρα δίνω πάλι το λόγο στην κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είμαστε λίγοι πια, είμαστε μεταξύ μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Μωράες, εξαιρετική δουλειά του, συγχαρητήρια μαζί με τους και εισηγητές βέβαια. Ε, πετύχατε μια συμφωνία μεταξύ Κομισιών, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, ε, όλοι βοήθησαν αυτός ο συμβασμός τον οποίο καταλήξαμε είναι ισορροπημένος και ευθυγραμμίζεται με την πρόταση του 2007. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογή στου δικαιούχου διεθνού προστασία θα εξασφαλίσει ψηλή, υψηλό επίπεδο προστασία και νομική ασφάλεια για του πρόσφυγε στην Ευρώπη και θα επιτρέψει την καλύτερη ενσωμάτωσή του στι κοινωνίε μα. Πρόκειται και για το ε, πρώτο ε, τούβλο ενός ε, πακέτου έξι νομοθετικών κειμένων είναι το πρώτο βήμα προς τον ε, στόχο μας να πετύχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου μέχρι το 2020, 12. Ε, ε, είναι σημαντικό που συμφωνούμε να κάνουμε αυτό το δύσκολο, δύσβατο αλλά απαραίτητο δρόμο προκειμένου να χτίσουμε αυτή την ενιαία πολιτική ασύλου. Σε ό,τι αφορά το θέμα των πινάκων συσχετισμού, το περιβόητο αυτό θέμα, η Κομισιόν έκανε μια δήλωση στο Συμβούλιο, να σας τη διαβάσω η Κομισιόν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή τη ε, να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν πίνακε συσχετισμού με τα μέτρα μεταγραφής ε, τα οποία θα έχουν ε, υιοθετήσει και να τα κοινοποιούν ε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη νομοθετική διαδικασία ε, με περισσότερη διαφάνεια και ε, να εγγυηθούν ότι οι εθνικές διατάξεις θα εφηγανίζονται με τις κοινοτικέ οδηγίες. Η Κομισιόν εκφράζει τη της για τον τρόπο με τον οποίο με, τα, με την υποχρεωτική σύσταση τέτοιων πινάκων μπορούμε να δεχτούμε ε, την υποκατάσταση αυτής της υποχρεωτικής ε, διάταξης ε, με ένα, με μια αιτιολογική σκέψη που θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προβούν στην κατάρτιση τέτοιων πινάκων, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προηγούμενο. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Κομισιόν θα προσπαθήσει να βρει μία ε, λύση σε αυτό το οριζόντιο θεσμικό πρόβλημα. Ελπίζω να συμφωνήσετε. Ε, το έχει καταγραφεί αυτή η δήλωσή μας ε, στα πρακτικά και απλώς την επανέλαβα. Σε ό,τι φορά αυτή την έκθεση είναι πολύ σημαντικό που καταλήξαμε συμφωνία και ξανά σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ερχόμαστε στους ομιλητές εν ονόματι των ομάδων. Πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Μαρία Νεντέλτσεβα για το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, θα ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κλόντ Μωράης για την εξαιρετική του εργασία και να τον ευχαριστήσω επίση για την ε, εξαιρετικό πνεύμα συνεργασία το οποίο έδειξε στι ε, σχέση με την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο. Κάναμε ένα άλμα προ τα εμπρό για ένα εναρμονισμένο σύστημα. Η συμφωνία που επιτύχαμε με το Συμβούλιο ήταν απαραίτητη και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μπορέσαμε να προχωρήσουμε με αυτόν τον με αυτό το ζήτημα. Το θέμα του ασύλου είναι φυσικά πολύ ευρύτερο, δεν θα πρέπει να παραιτηθούμε. Θα είναι απαραίτητο να υπάρξει περαιτέρω διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. αυτά ήθελα να πω ω εισαγωγή. Έμπει τη ουσία, λοιπόν, έχω δίχω να επαναλάβω τον εισηγητή, να επανέλθω σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα να τονίσω την σημασία τη ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στι χώρε μα. Οι κοινωνίε μα, οι μετανάστε αποτελούν ένα θετικό ατού για τις ε, χώρες μας, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οτιδήποτε κάτω από οποιασδήποτε ε, προϋποθέσεις ε, διακόπτει ο Πρόεδρος την ομιλήτρια ζώντας να επιβραδύνει τον ρυθμό ομιλίας. Έχουμε άτομα τα οποία εργάζονται εδώ και 5-10 χρόνια στην Ευρώπη και δεν καταφέρνουν να γνωρίσουν την γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας. Πώς μπορούν τα πρόσωπα αυτά να δραστηριοποιηθούν στις κοινωνίες πώς ε, μπορούμε παράλληλα να ε, ξεπεράσουμε τον, ε, αυτά τα εμπόδια, αυτούς τους φραγμούς πρέπει να υπάρξει εκμάθηση της γλώσσας διότι μέσω της γλώσσας μπορούμε να αποκτήσουμε η γνώση και της κοινωνίας, του πολιτισμού της χώρας κλπ. Και εδώ αναφέρω την απογοήτευσή μου διότι το Συμβούλιο αρνήθηκε να συμπεριλάβει τις πινέκες αντιστοιχίες στο κείμενο. Φυσικά δεν μπορούμε να να σταματήσουμε τις συζητήσεις λόγω αυτού του γεγονότος, αλλά αναρωτώ μεθά πότε το Συμβούλιο θα επιτρέψει την διάδοση προφοριών των απαραίτητων που είναι ε, που αφορούν την εφαρμογή των οδηγιών από τα κράτη-μέλη. Διότι αναρωτώμεθα εάν η Κομισιόν δεν μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο τα κείμενα πραγματικά μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία, τι συμφέρον έχουμε στο να νομοθετούμε. Και επί του θέματος αυτού θα να συγχαρώ την κυρία Επίτροπε για την δήλωση που έκανε και μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα, διστήσω, θα δώσω μάλλον το λόγο στη κυρία Σεσίλοβο Βίλκστρομ διότι η κυρία Φλασίκοβα απουσιάζει. Εξ των φιλελευθέρων δημοκρατών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν επιθυμώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Κλοντ Μωράης, που ως συνήθω έκανε μια εξαιρετική και πολύ σοβαρή εργασία. Και που θα ήθελα να πω ότι Πολλά από αυτά τα άτομα μένουν για μεγάλο διάστημα ή και για ολόκληρο τον βίο τους, διότι πολλά από αυτά τα πρόσωπα διώκονται στις χώρες τους και ε, τα πρόσωπα τα οποία τυχάνουν διεθνούς ε, προστασίας χρειάζεται να ε, θεωρηθούν ως ε, μονίμως διαμένοντα μετά από μια πενταετία. Αλλά το Συμβούλιο έχει διαφορετική άποψη από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Και αυτό με απογοητεύει ιδιαίτερος. Επίσης να αναφερθώ στο ζήτημα της οικογένειας η οποία θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ζήσει ενωμένη. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να εγκρίνει την ε, έκθεση. Λυπάμαι που το Συμβούλιο δεν δέχθηκε τους πίνακες ανησυχίας. Αλλά φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επανέλθει με την οδηγία περί ασύλου. Έχουμε κάποιες προθεσμίες ε, που θα πρέπει να τηρήσουμε, π.χ. το 2012. Δεν θα πρέπει λοιπόν να, να παραμείνουμε στις θέσεις μας, αλλά χρειάζεται να υπάρξει μια κοινή θέση σε ό,τι αφορά το ζήτημα ασύλου. Διαφορετικά ο όρος αλληλεγγύη θα κενωθεί από το περιεχόμενο του. Ευχαριστώ τον κύριο Μωράς για την εργασίες του, αλλά και για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ και εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και να δώσω το λόγο τώρα εξ των Πρασίνων την κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή Λίμπε μετέβη στην ε, Αθήνα και συζήτησα με τον Μαμούτ, ο οποίος είναι 26 ετών και έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ελλάδας και έπειτα μετέβη στην Σκάτοχώρες ε, να, προτιμούσε να παραμείνει στις Σκάτοχώρες αλλά τελικά τον ε, επαναπρόθεσαν στην Ελλάδα. Και όταν θα αποκτήσει το καθεστώς του ετούνους ασύλου στην Ελλάδα, δεν θα μπορέσει να κυκλοφορήσει ελεύθερος και θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Και υπάρχουν χιλιάδες άτομα στη, όπως, στη θέση συγγνώμη, του Μαμούτου και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα χέρια του και να τροποποιήσει τα την κατάσταση και ο συνάδελφος Κλοντ Μωράης ανέλαβε αυτό το νέο διάβημα. Διότι ο Μαμούτ θα είχε προτιμήσει να παραμείνει στις κατοχώρες όπου είχε γνωστούς αλλά θα χρειαζόταν ε, να εφαρμοστούν οι πίνακες. αντιστοιχεία στην περίπτωση αυτή, διότι ο Μαμούτ είχε δικαίωμα να γνωρίζει πώς ε, θα εφαρμοζόταν παρόμοια οδηγία στις κάτω χώρες στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Μωράης, ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και για το καλό του Μαμούτ και όλων των υπολείπων. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε μία λύση. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους και ε, πρωτίστως τον κύριο Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή. Συμφωνώ πλήρως με την έκθεση. Νομίζω ότι χορηγεί καινούργια δικαιώματα σε όσοι ετούνται διεθνή προστασία συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων τους ε, εγγυάται δικαιώματα τα οποία αποδίδουμε σε ανθρώπους που έρχονται από τρίτες ε, χώρες και έχουν ζήσει για πάνω από πέντε χρόνια στις, ε, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα. εγώ προέρχομαι από μια χώρα που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα Πρέπει κανεί να περιμένει πέντε χρόνια για να αποκτήσει το δικαίωμα που δίνει αυτή η νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, Ιδιαίτερο για μια χώρα η οποία δέχεται ένα τεράστιο αριθμό ε, ατόμων που έρχονται και μπλοκάρονται σε μας. Ε, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. Το είδαμε πρόσφατα αυτό, ε, από κοντά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρειάζεται να περιμένουν πέντε χρόνια για να καταφέρουν ε, να αποκτήσουν αυτά τα δικαιώματα για τα οποία συζητούμε. Το καθεστώς δηλαδή του επιμακρών διαμένοντος και που τους δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η πιο γρήγορη χρήση αυτού του δικαιώματος θα βοηθούσε μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα. Για να γίνει ακόμα καλύτερη λοιπόν αυτή η νομοθεσία, αυτό το νομοθετικό κείμενο, θα έπρεπε ε, αυτά τα άτομα να μην χρειάζεται να περιμένουν πέντε χρόνια για να αποκτήσουν αυτή την άδεια, αυτό το καθεστώς. Θα ήθελα παρόλα αυτά να ευχαριστήσω τον κύριο Μωράη που το αναγνώρισε και έκανε ό,τι μπορούσε για να το συμπεριλάβει έστω και συμβολικά στην ε, εξήγησή του. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γιώχαν Εντσιού που εκπροσωπεί τη Ρουμανία. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον, τον κύριο Μωράης. να τον ευχαριστήσω για τις προσπάθειες ε, που καταβάλει κάθε φορά που είναι συντονιστής ε, στο, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η οδηγία αυτή καλύπτει ένα νομικό κενό, επιτέλους. Στο θέμα των, των δικαιωμάτων διαμονής, καλύπτει δηλαδή πλέον τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας άτομα τα οποία διαμένουν σε ένα κράτος μέλος και που βρίσκονται ε, σε μια επισφαλή νομική θέση και κατάσταση διότι προς το παρόν δεν χαίρουν ε, το, του καθεστώτος ε, επιμακρών διαμένοντος όπως άλλοι πολίτες. Η χορήγηση του καθεστώς αυτού σε αυτά τα άτομα θα πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις υπό τον όρο ότι έχουν διαμείνει για μία χρονική περίοδο προκαθορισμένοι όπως και οι υπόλοιποι. Θα πρέπει να λαμβάνετε μάλιστα υπόψη το σύνολο της διαμονής αυτών των ατόμων σε, στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που υπέβαλαν αίτηση για την άδεια διαμονής. Αυτά τα άτομα ε, είναι ευάλωτα όσο είναι στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο η άρση του ε, δικαιώματος διεθνούς προστασίας, η, άρση της, η, ακύρωση της άδειας διαμονής θα πρέπει να υπόκειται ε, στο, στους όρους του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Πιστεύω θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση του κ. Μωράες είναι ένα τμήμα του γενικού πακέτου ρύθμιση του συστήματο ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουλευτά. Τώρα θα δώσω... Ε, πέρασουμε μάλλον τη διαδικασία κάτσου διάει. Έχουμε μόνο έναν αγορητή, ο κύριος Όμπερ Μάιερ. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν βλέπω τόσο αισιόδοξα αυτό, αυτή την έκθεση αλλά ανησυχώ για τους πολίτες μας διότι ε, εάν κάποιος ε, επιτύχει το καθεστώς οπιμεκρών διαμένοντος θα παραμείνει εις ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου επιθυμεί και θα κοιτάξει να βρει ε, τη χώρα όπου υπάρχουν ε, πολύ υψηλότερες ε, κοινωνικές προϋποθέσεις, πολύ καλύτερες και μπορεί να καθυστερήσει η διαδικασία πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν τα κράτη που έχουν υψηλό βαθμό κοινωνικής προστασίας και θα υπάρχει μεγάλη καλύτερη προσέλευση προσφύγων και ως εκ τούτου εγώ θα καταψηφίσω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ και έτσι Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει αυτή την συζήτηση και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω πολλά να σας πω κυρία, κύριε Πρόεδρε διότι απλούστατα έχω μία έκκληση προς τον κύριο Μωράης και στους άλλους ότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα και ελπίζω ότι θα υπάρχει ε, ισχυρή στήριξη αύριο διότι είναι η το πρώτο βήμα για το πακέτο του ασύλου για το 2012. Βασίζομαι λοιπόν στην συνεργασία σας για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε και τα επόμενα νομοθετήματα. Ευχαριστώ κυρία, κυρία Επίτροπε και τώρα δίνω το λόγο στον εισηγητή κύριο Μωράες. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Επίτροπε. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν καταφέραμε να κάνουμε το πρώτο βήμα για να το ολοκληρώσουμε για το άσυλο, ελπίζω ότι θα επιτευχθεί αύριο, είναι διότι επειδή το άσυλο παραμένει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα σε αυτό το κοινοβούλιο, όπως εξέγησε ο κύριος Μπουσουτή, ο οποίος είπε πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα, ιδίως για τις μικρές χώρες, όπου το άσυλο μπορεί να έχει υπορμεγέθη επιπτώσεις πέραν των συνόρων των δεδομένων χωρών. Γι' αυτό παρόλο που στο επεξηγηματικό υπόμνημα θα ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν ε, ε, ε, υπάρξουν ορισμένες ρυθμίσεις όσον αφορά τις απελάσεις πιστεύω ότι όλα τα θέματα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα πάνε καλά και το, θα μας συνδράμει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Σαρζεντίνη, ήθελα και εγώ να σας πω ότι βεβαίως είναι σημαντική η και συσχετισμού, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να περιμένουμε για να εφαρμόσουμε το άσυλο να εφαρμοστούν οι πίνακες συσχετισμού. Ελπίζω όμως ότι ακούει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την βοήθειά τους και την πρόθεση αυτής της εκθέσεως μετά από τόσο χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα σας ανακοινώσω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος αυτό και θα έχουμε την ψηφοφορία αύριο το μεσημέρι. Τώρα φτάνουμε ε, στην κοινή συζήτηση για το θέμα της περιφερειακής πολιτικής. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω ε,